Okay, wir fahren kurz So now we will start with our next item. Και τώρα πάμε στο επόμενο θέμα της μέσης διάδεξης που είναι οι ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εδώ τον Επίτροπο Σπίτλο. Η πρώτη ερώτηση για αυτόν προέρχεται από την κυρία Τεγκαροπούλου Κράτσα. Το θέμα είναι η συμμετοχή των γυναικών στις ευθύνες αγορά εργασία. είναι εδώ κυρία Κράτσα, κύριε Επίτροπο έχετε το λόγο. Εδώ είναι μάλλον κυρία Κράτσα. Αλλά ο κύριο Επίτροπο έχει το λόγο. Πρόεδρε, ο αριθμός των γυναικών που έχουν θέσεις ευθύνης έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και όμως παρόλα αυτά θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι τα ενία σε όλες αυτές τις θέσεις στη δουλειά και στην πολιτική θα κρατούν οι άντρες. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη ισορροπία. Όπως θα πρέπει να βρεθεί και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και επιγενικού βίου, ώστε να μπορέσουμε να άρουμε τους φραγμούς που βρίσκουν γυναίκε στον δρόμο του, ούτω ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν για αυτέ τι θέσει υπεύθυνε. Στην τελευταία δεκαετία πάντω σημειώθηκε μια πρόοδο στι περισσότερε χώρε τη Ένωση. Πάντω οι αλλαγέ επέρχονται σιγά σιγά. Και ακόμα δεν έχουν πάρα πολλέ γυναίκε σε σημαντικέ θέσει διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και ιδίω στι ε, επιχειρήσεις. 9 στου 10 όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, 9 στα 10 εκτελεστικά στελέχη, οι μέλη τέλο πάντων ιδιωτικών συμβουλίων είναι άντρε και μόνο 3% είναι. 3% των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχουν ένα διοικητικό συμβούλιο του οποίου πρόεδρος είναι γυναίκα. Πιστεύουμε στα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η κατάσταση επιδέχεται βελτίωσε, ανάλυση, σύγκριση των ε, δεδομένων, ε, να εκμεταλλευτούμε τα δίκτυα και την υπάρχουσα εμπειρία. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που υποστηρίζει τις γυναίκες. Αυτό το συγκροτήσαμε τον Ιούνιο του 2008 εμείς. Και έτσι μπορούμε να προωθήσουμε κάποια μέτρα που θα βοηθήσουν δίκτυα λοιπόν των γυναικών. Να γίνει συνειδητοποίηση του προβλήματο, να ενθαρρυνθούν οι γυναίκε τελικά να μπορέσουν να επιδιώξουν την κατάληψη ανωτέρων θέσεων. Θα θέλουμε με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι αρκετά κρατημέλη έχουν λάβει πρωτοβουλίες όπως ε, τον επισημένο το πρόβλημα στον ιδιωτικό τομέα, ε, κατάρτιση των γυναικών που θέλουν ε, να ξεπεράσουν αυτούς τους φραγμούς, να κατράβουν υπευθύνες θέσεις. Επίσης, γίνεται προσπάθεια να υπάρχει ένα σύστημα ανταμοιβής των ε, επιχειρήσεων που επιδιώκουν περισσότερο ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Με μεγάλο ενδιαφέρον επομένω παρακολουθούμε κυρίω το νορβηγικό μοντέλο. Βέβαια κάθε χώρα θα πρέπει να υιοθετήσει ό,τι τη πάει περισσότερο. Άρθρο 141 παράγραφο 4 τη συνθήκη, αποτελεί μια αφετηρία ούτω ώστε τα κρατημέλη να πάρουν κάποια θετικά μέτρα. Πάντως υπάρχει νομολογία περιοριστική από το 10. Σύμφωνα με το 10 δεν είναι δυνατόν να ληφθούν αυτοδικαίω αυτομάτω κάποια μέτρα. Θα πρέπει τα μέτρα να θεσπίζονται αναπερίπτωση. 2010 θα φτιάξουμε μια στατική κατευθυντήριες γραμμές, θα κάνουμε μια μελέτη των επιπτώσεων, θα προβούμε και σε μια ανάλυση του τι έχει γίνει από το 2006 και μετά. Ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε κάποιε θέσει υπεύθυνε. Αυτό θα είναι προτεραιότητά μα. αρχάς του επομένου έτους θα ξεκινήσει αυτή η καινούργια στρατηγική για ανάπτυξη κλπ. Ούτω ώστε να μπορέσουμε σε αυτή τη νέα στρατηγική να έχουμε ω επίκεντρο την ισότητα ανδρών και γυναικών. Και σα τονίσω, εδώ δεν είναι θέμα πολιτικό, δεν είναι θέμα ηθικό. Η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι θέμα οικονομικό. Εάν η κοινωνία δεν καταφέρει να εκμεταλλευτεί τι δεξιότητε, τις δυνατότητε όλε που υπάρχουν στι γυναίκες, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει με επιτυχία στο μέλλον. Γι' αυτό σας λέω, κυρίε και κύριοι, θα πρέπει κανείς να δεσμευτεί χωρίς κανένα περιορισμό ή στο να προσπαθήσουμε οι γυναίκες να καταλάβουν και αυτές κορυφαίε ε, θέσεις σε μια φιλόδοξη Ευρώπη. Κύριε Κράτζα. Έχετε Κύριε Επίτροπε, άλλη μια φορά για τη δέσμευσή σα υπέρ τη προώθηση των γυναικών σε θέσει ευθύνη. Επιτρέψτε μου να σα πω ότι ήταν πιο συγκεκριμένο το ερώτημά μου. Εν ώψη τη αναθεώρηση ε, των στόχων τη Λισαβόνα και τη αξιολόγηση του χάρτη πορεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του ελλείμματο των γυναικών σε θέσει ευθύνη στην αγορά εργασίας. το μοντέλο το νορβηγικό στο οποίο αναφερθήκατε θα αποτελέσει μια έμπνευση μιας κατευθυντήριας γραμμής ε, και η νομολογία του δεκ που είπατε πώς συνδέεται με αυτό είναι ενθαρρυντική ή αποθαρρυντική για να πάρετε μια θέση. σας ευχαριστώ πολύ. μια θέση ως ευρωπαϊκή επιτροπή υπέρ μια κατεύθυνση. ευχαριστώ. ευχαριστώ. E, e, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφή στα όσα είπα. σω όμως θα πρέπει να είμαι ακόμη πιο σαφή. Οι ίσες ευκαιρίε είναι ήδη στο επίκεντρο της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι άποψη της Επιτροπής Ανεξάρτητα Οικονομικές και Ηθικές Απόψεις. Η ισότητα των ευκαιριών θα τονιστεί, θα υπογραμμιστεί στις μελλοντικές στρατηγικές και θα προτείνουμε σε όλα τα κατάλληλα έγγραφα τα απαιτούμενα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε επιτυχία στον τομέα αυτό. Βεβαίως, πάντοτε θα πρέπει να παραμένουμε μέσα στα όρια και τους περιορισμούς της συνθήκης, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε ε, περισσότερο τα μέσα ε, της συνθήκης. Ο κύριος Λάρξη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Πολύ ωραία ήταν αυτά που μας είπατε, όμως ε, θα πρέπει να δούμε και να έχετε κατά το εξής. Ε, όταν είναι κανείς πολιτικός πρέπει να γνωρίζει και τι έχει πράξει. Τα τελευταία λοιπόν πέντε χρόνια, εκείνο το οποίο βιώσαμε, σε εσά τουλάχιστον, είναι ότι εσείς συνεργάζεστε μόνο με άνδρες. Και πώς είναι δυνατόν η Κομισιόν να μην έχει ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων. Και από ό,τι φαίνεται ούτε και στο μέλλον δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Μήπως λοιπόν θα ήταν σκόπιμο η Κομισιόν να δώσει το καλό παράδειγμα έτσι ώστε μετά να ληφθούν και άλλα ε, παρεμφερή μέτρα. Ναι, ναι, βεβαίως. Αξίζει να τονίσουμε ότι η Επιτροπή αυτή είναι μια Επιτροπή που έχει σπάσει ρεκόρ ε, από την άποψη του αριθμού των γυναικών επιτρόπων. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι οι συνάδελφοί μου γυναίκες έχουν ε, τα βασικά χαρτοφυλάκια. Η Νέλη Κρούς, Ντάρια Γκριμπεσκα και, και οι κυρίες επίτροποι έχουν ε, χαρτοφυλάκια κλειδιά. Η Επιτροπή λοιπόν είναι μια, ένας παραδειγματικός θεσμός η επιλογή βεβαίως ε, υποψηφίων γυναικών για τη θέση των επιτρόπων είναι έργο, είναι ευθύνη και καθήκον των κρατών. Θα πρέπει τα κράτη να διαλέξουν γυναίκες για επιτρόπους και η Επιτροπή η σύνθεσή της θα αντανακλά αυτές τις επιθυμίες των κρατών. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στο σύνολό της θα, θα έχει αλλαγές, διότι έχουμε αναγνωρίσει ότι δεν έχουμε ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Χαίρομαι όμως, διότι χάρη ε, στις ε, προσπάθειες του συναδέλφου Σιμ Κάλλας αν συγκρίνετε τους αριθμούς της αρχής και τους αριθμούς που έχουμε τώρα τα στοιχεία θα δείτε ότι έχουμε κάνει σημαντικές πρόοδους αλλά έχετε δίκιο έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε σε μια ικανοποιητική κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση. Έχω ένα σχόλιο για αυτή την ερώτηση με ε, εκπλήσει αυτή η συζήτηση που έχουμε κάθε χρόνο και βλέπω ότι η πολιτική πρέπει να αλλάξει αν θέλουμε πολύ περισσότερα άτομα να εμπλέκονται, να συμμετέχουν και πολύ περισσότερες γυναίκες στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Ε, εμείς όπως η λειτουργία μας ως Κοινοβουλίου δεν το ευνοεί αυτό. Είμαστε, ε, έχουμε παιδιά, αγόρια και κορίτσια και πρέπει να το κάνουμε. Έχω, έχω κάνω αυτή τη διαδρομή, αλλά έχω κάποιον που μένει στο σπίτι. Πρέπει λοιπόν να, έχουμε, είμαστε πρακτικοί ως προς το θέμα αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπος ίσως. Ναι. Στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις επεσήμανα ότι υπάρχει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη σειρά καταστάσεων, μερικές καταστάσεις θετικές, μερικές λιγότερο θετικές. Σαφώς, τελικά, κάθε άτομο, κάθε ανθρώπινο όν αποφασίζει για τον εαυτό του. Βεβαίω, ορισμένα θεσμικά όργανα, ορισμένοι οργανισμοί, ορισμένες πολιτικέ, ορισμένε διευθετήσει επιτρέπουν στα άτομα μεγαλύτερη ελευθερία από ό,τι άλλε. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι προφανές ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να επιτύχουμε ίσες ευκαιρίες, ισότητα ευκαιριών. Ε, θα πρέπει να εξαλείψουμε κάθε διάκριση, άμεση έμεση διότι για την ώρα όλοι, όλες οι γυναίκες δεν έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα που έχουν οι άνδρες όσον αφορά στη λήψη των αποφάσεων. Κυρίως όσον αφορά στην ε, πρόσβαση σε πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Έχουμε τώρα μια ερώτηση από τον κύριο Τζάκι Ενά, αλλά φοβούμε ότι θα πρέπει να αναβάλουμε ε, αυτήν την ερώτηση, να την παραλείψουμε, ε, διότι είναι απόν ο ερωτών. Το ίδιο ισχύει και για την Σεσίλια Βίλτστρομ, η οποία δεν είναι παρούσα εδώ στην αίθουσα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Σπίτλα για το χρόνο του και για τις απαντήσεις του και βλέπω τον Επίτροπο Ορμπάν, ο οποίος έρχεται να λάβει θέση. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον Επίτροπο Ορμπάν να καθίσει. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Αυτή είναι μια ερώτηση του κυρίου Πόσελτ, ο οποίος παρίσταται στην αίθουσα και πρόκειται για την εκμάθηση γλωσσών στις παραμεθόριες περιοχές. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Κοιτάξτε, εφόσον είμαι ο Επίτροπος Αρμόδιο για την πολυγλωσσία, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Στο άρθρο 149 στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και της οργάνωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών. Όπως ε, αναφέρεται λοιπόν ε, στο προαναφερθέν άρθρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια στο να ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και εφόσον κρίνεται απαραίτητο να στηρίζει τις ε, δράσεις των ε, κρατών μελών ε, στον τομέα αυτό. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η επιλογή των γλωσσών που διδάσκονται στα σχολεία των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη την ε, γεωγραφική κατανομή αλλά και την παρουσία εθνικών μειονοτήτων. Αυτό λοιπόν αναφέρεται στην ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου του 2008 που φέρει τον τίτλο ε, «Πολυγλωσσία στην Ευρώπη. Κοινή δέσμευση». Η ανακοίνωση αυτή επισημαίνει το γεγονός ότι ε, πρέπει να καταβάλουμε και άλλες προσπάθειες έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των γλωσσών που διδάσκονται κυρίως όσον αφορά την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας ε, κυρίως εκεί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες που επικρατούν. Όσον αφορά την επέκταση αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή το πόσε γλώσσε ε, θα μπορούν να διδάσκονται ως ε, δεύτερη επιλογή, εμείς προτείνουμε την επικοινωνία ανάμεσα στους άμεσους ενδιαφερόμενους και αυτό να στηρίζεται από το πρόγραμμα Comenius Regio, η συνεργασία με τους άμεσα ενδιαφερόμενους ε, επιτόπου, όπως σας είπα, είναι κάτι που πρέπει να προωθηθεί, όπως και η αδελφοποίηση με άλλες χώρες τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζει την εκμάθηση όλων των γλωσσών που ομιλούνται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των γλωσσών των μειονοτήτων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει την ε, μετακίνηση και πέρα από τα σύνορα, έτσι ώστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να μάθουν νέες γλώσσες η το πρόγραμμα ε, συνεργασίας ε, και πέρα από τα σύνορα, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να στηρίξει και άλλες δραστηριότητες ε, για την εκπαίδευση των νέων, την, την κοινωνική συμπερίληψη των νέων και εδώ παίζει ρόλο και η γλώσσα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, Educative Command, το οποίο στηρίζεται από το διασυνορικό πρόγραμμα ε, Γαλλίας και Αγγλίας ε, για την περίοδο 2007-2014. Εκεί στόχος είναι να υπάρχει ένα διασυνοριακό μάλλον υπερεθνικό δίκτυο σχολείων, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να μάθει κανείς ξένες γλώσσες και να είναι δυνατόν να προσφέρονται πληροφορίες ε, σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δις ε, ευρώ. Άμεσα ενδιαφερόμενοι ε, μπορούν να βρίσκονται και στις δύο πλευρές της μάχης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένα πρόγραμμα από ένα διαφορετικό μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει συμπεριληφθεί σε τρία υπερεθνικά προγράμματα ε, πρόκειται το πρόγραμμα Αυστρίας-Τσεχίας, Αυστρίας-Σλοβακίας και Αυστρίας-Ουγγαρίας. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους νέους για υπερεθνικές δραστηριότητες στο κέντρο της ε, Ευρώπης προσφέροντάς τους εκπαίδευση και βοηθώντας τους να αποκτήσουν γλώσ... ικανότητες γλώσσας και ε, γνώσεις επικοινωνίας. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 791.000 ευρώ. Τώρα, θέλετε ε, κύριε Πόσελτ να υποβάλλετε μία συμπληρωματική ερώτηση. Ο κύριος Πόσελτ, Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Να, ειδού το παράδειγμα. Εσεί είστε το παράδειγμα για την πολυγλωσία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Επίτροπο το εξή. Πρώτον, κατά πόσον το πρόγραμμα το οποίο ανέφερε Αυστρία-Ουγγαρία και Αυστρία, Τσεχία και Αυστρία, Σλοβακία, κατά πόσον ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να ελοπιθεί και ανάμεσα στην Ουγγαρία και τη, και Σλοβακία. Πολιτικά αυτό θα ήταν πολύ ε, χρήσιμο. Δεύτερον, θεωρώ ότι πράγματι στι παραμεθόριε περιοχέ πρέπει κανεί να μαθαίνει καλύτερα τη γλώσσα τη γειτονική χώρα, να μαθαίνουν οι Αυστριακοί περισσότερα Ουγγρικά και Τσεχικά. Ε, Βεβαίω ε, και στα νηπιαγωγεία και εμένα όμως με ενδιαφέρει κυρίως ε, η εκπαίδευση των ενηλίκων, η διαβίου μάθηση, οι πιο ηλικιωμένοι να έχουν περισσότερες δυνατότητες να μαθαίνουν τη γλώσσα της γειτονικής χώρας. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη συμπληρωματική ερώτηση. Ο κύριος Επίτροπος έχει το λόγο. Σας ε, ευχαριστώ για αυτή τη συμπληρωματική ερώτηση. Εις ό,τι αφορά το πρώτο θέμα που αναφέρατε, θα είχα να πω το εξή. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα πρόγραμμα ε, μεταξύ Ουγγαρίας και Σλοβακίας. Είμαστε απολύτως πρόθυμοι να εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο για να συνεισφέρουμε στην εξέβρεση αμοιβαία αποδεκτών και από τις δύο χώρες λύσεων. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέμα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία για την ε, ταχεία και έγκαιρη εκμάθηση ξένων γλωσσών. Έχει ήδη αποδειχθεί καρποφόρα και συνδυάζεται και με την πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει ε, ενώπιον των γονέων να ενθαρρύνουν τα μικρά παιδιά τους ηλικίας 2-6 ετών να ξεκινήσουν την εκμάθηση ξένων γλώσσων. Εις ό,τι αφορά το δεύτερο σας ερώτημα, τη διαβίου μάθηση. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της πολιτικής που ακολουθούμε. Έχουμε πολλά προγράμματα με στόχο ακριβώς αυτόν, την εκμάθηση των ξένων γλωσσών που διευκολύνουν τις πολιτισμικές και διαπολιτισμικές επαφές. Κυρίως για αυτούς που είναι εκτός του κλασικού εκπαιδευτικού συστήματος. Για τους μειονεκτούντες, για τους συνταξιούχους, για τους άνεργους. Και βεβαίως χρηματοδοτούμε αυτά τα προγράμματα. Κάτι το οποίο έχει και αυτό σημασία γιατί συνάδει με την στρατηγική που ενέκρινε το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε όλοι οι πολίτες, όχι μοναχά οι νέοι να έχουν δυνατότητα να μάθουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες. E, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τις ενδιαφέρουσες αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε. Απαντώντας όμως στο ερώτημα, ο Επίτροπος ε, ανέφερε έστω και εν παρόδο τα σχολεία. Εντάξει, καλώς. Υπάρχουν όμως και πανεπιστήμια που είναι μάλιστα σε παραμεθόριες περιοχές όπως το Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Τα χρήματα που αναφέρατε ότι είναι διαθέσιμα κύριε Επίτροπε μπορούν να διατεθούν και προς ε, μεθοριακά, ε, παραμεθόρια συγγνώμη, πανεπιστήμια. Εγώ στο βαθμό που τα πανεπιστήμια είναι σε θέση να υποβάλλουν προγράμματα που να είναι επιλέξιμα, να πληρούν δηλαδή τα κριτήρια του προγράμματος διαβίου μάθησης για την περίοδο 2007-2013, γιατί σε αυτή βρισκόμαστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απολύτως διατεθειμένη μετά την διαδικασία επιλογής βεβαίως να τα χρηματοδοτήσει. Υπάρχει δε μια σειρά προγραμμάτων που ήδη χρηματοδοτούνται υπό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που έχουν ως εταίρους ένα πολύ σημαντικό αριθμό πανεπιστημίων που προέρχονται απανταχού της ενώσεως. Η απάντησή μου λοιπόν καταφατική. Ναι, αυτό το οποίο δεν μετράει περισσότερο είναι η ποιότητα του φακελού που παρουσιάζουν οι υποψήφοι. Κύριε Ρούμπιχ, είναι... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το δικό μου το ερώτημα αφορά το εξή. Έχουμε πολλά προγράμματα έρασμος για του ε, φοιτητέ. Έχουμε προγράμματα για νέου επιχειρηματίε. Τώρα κάτι καινούριο. Έχουμε και προγράμματα για δημοσιογράφου. Πιστεύετε εσεί ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προγράμματα έρασμος για να βελτιώσουμε την επικοινωνία στι παραμεθόρες περιοχέ και αν το εγκρίνετε αυτό, πού ακριβώ θα αποδίδατε το βάρο. Ευχαριστώ. Uh, răspunsul Η απάντηση είναι καταφατική. Διότι το έρασμος είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πριν από περίπου μία εικοσαετία το βλέπει ο κόσμος με επιφυλάξεις. Τώρα όμως είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης. Ε, πήγα πολλές φορές και σε πρωτεύουσα κρατών μελών, αλλά και στην επαρχία. Και έτσι μπόρεσα να δω πόσο θετικά αποτελέσματα έχει αυτό το πρόγραμμα. Κάποιος ανέφερε πριν το θέμα των πανεπιστημίων σε Πολωνία και Γερμανία. Θυμάμαι ότι όταν επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας διαπίστωσα ο ίδιος πόσοι Γερμανοί φοιτητέ φοιτούσαν εκεί μέσω του έρασμους. Έτσι ήταν δυνατόν να μάθουν και τα πολωνικά αλλά και την κουλτούρα, τον πολιτισμού της χώρας. Αυτό σας δείχνει Πόσο αποτελεσματικό είναι το πρόγραμμα. Με κατακλείτη, σας υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος κ. Μπαρόσο το είπε ότι δηλαδή πρώτη θέμεθα στο άμεσο μέλλον να αναλάβουμε πρωτοβουλίε στοχευμένες ούτως ώστε να βελτιωθεί η κινητικότητα των νέων και έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλες τις δεξιότητες που χρειάζονται, όλο ένα και περισσότερο. Ο πρώτος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τι ήρθατε να μας δείτε, για το χρόνο μας διαθέσατε, για όλα μας είπατε. μέσα στα Ρουμάνικα. Καλά Και τώρα ο κύριος Κάλλας. Η επόμενη ερώτησή μας είναι από τον κύριο Νικόλαο Χουντή και το θέμα είναι ολιγορία της Επιτροπής στην ε, διερεύνηση του σκανδάλου της Siemens. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στα θέματα διαφθοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά πρέπει να πω ότι όσον αφορά στο σκάνδαλο της Siemens και όλα τα θέματα γύρω από τη Siemens και ε, τα θέματα που αφορούν άμεσα ή έμεσα τη Siemens ε, είναι, ε, είναι με πολλά. Και τα θέματα, τα, η Όλαφ ασχολήθηκε τον δεύτερο τρίμηνο σχετικά με το θέμα αυτό και υπάρχει μια δικαστική, ε, δικαστικά, ε, το δικα, δικαιοσύνη ασχολείται με το θέμα αυτό στην Γερμανία και η Όλαφ παρακολουθεί το θέμα στην χώρα αυτή. Δεύτερον, ε, περίπτωση της Όλαφ σχετικά με έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρακολουθούνται, εξετάζονται από την Όλαφ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης, ε, που χρηματοδοτούνται από ε, ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αξιολογούνται επίση από την Όλαφ ούτω ώστε να προσδιοριστεί αν υπάρχουν, υποψίε σοβαρέ υποψίες σοβαρές απάτης σχετικά που ευνοούν ορισμένα χρηματικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνα, η Όλαφ θα αποφασίσει αν θα υπάρξει προσφυγή σχετικά με την υπόθεση αυτή. Επίσης ε, τέταρτη υπόθεση στην ε, Ισπανία έχουμε την απόφαση ε, σχετικά με διαρθρωτικά ταμεία όπου η Siemens είχε εμπλακεί. Οι εθνικές αρχές στη δεκαετία του 90 ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και οι δικαστικές διαδικασίες έκλεισαν και από την Όλαφ. Επίσης ε, κατηγορήθηκαν πάρα πολύ για απάτη ε, και υπήρξαν φυλακίσεις και πρόστιμα που επιβλήθηκαν. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε αυτήν την περίπτωση η Siemens αθώθηκε στην, ε, στην πρωτόδικη απόφαση της 20 Ιουνίου 2006 του πρωτοδικίου της Ισπανίας. Η γενική εικόνα λοιπόν όπως με όλες αυτές τις περιπτώσεις Βεβαίως ε, η Όλαφ ε, δεν είναι ιδιοκτική αρχή. Η Όλαφ ε, περιλαμβάνει τα κράτη τα οποία πρέπει να ενημερώνουν την Όλαφ και η Όλαφ να παρακολουθεί τα θέματα στα οποία χρησιμοποιούνται πόροι ευρωπαϊκοί, πόροι κοινοτικοί. Ερευνώνται όλα αυτά τα θέματα. Αυτή είναι η γενική εικόνα και η Όλαφ επίσης συμμετέχει ε, σε θέματα διεθνούς συνεργασίας και συνεργάζεται με άλλους διεθνείς οργανισμούς για την καταπολέμηση της ε, κακής χρήσης χρημάτων που διατίθεται ε, για βοήθεια και για έργα σε σχέση με ορισμένα στοιχεία συγκεκριμένων υποθέσεων. Αν το αξιότιμο μέλος έχει συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα ήταν χρήσιμα, θα μπορούσε να τα υποβάλει στην Όλαφ η οποία θα τα αξιολογήσει και θα λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις σύμφωνα με την εντολή της Όλαφ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Χουντή έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η αίσθηση στην ελλάδα για το σκάνδαλο siemens είναι αυτό που γράφτηκε χαρακτηριστικά στον τύπο. ότι το σκάνδαλο το μεγαλύτερο στην ε, μεταπολεμική ελλάδα βαδίζει οριστικά για τη διαγραφή του μετά από την δεύτερη απόφαση του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου τη Γερμανία, το οποίο αναφέρει ότι ο κύριος χριστοφοράκος πρώην διευθυντή τη siemens ελλάς και αρχιερέα τη διαφθορά, δεν μπορεί να εκδοθεί από τη γερμανία στην ελλάδα. αυτή είναι η αίσθηση. έτσι εξελίσσεται στην ελλάδα το σκάνδαλο που με βάση ομολογίες και καταδικαστικές αποφάσεις γερμανικών δικαστηρίων έχουν και ενέχονται κρατικοί λειτουργοί οι οποίοι επί σειρά ετών δωροδοκούνταν για να αναθέσουν άγνωστον αριθμό προμηθειών και έργων που απολάμβανε οι ζήμες με το μαύρο χρήμα που διακινούσε. Ξαναρωτάω κύριε Επίτροπε, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι οι περισσότερες από αυτές οι προμήθειες είναι συγχρηματοδοτούμενα έργα μόνο οι υπηρεσίε σα και δυστυχώ σήμερα η απάντησή σα το ίδιο επιβεβαιώνει προσποιούνται ότι δεν το γνωρίζουν οχυρωμένε κατά την άποψή μου σε αυθαίρετε διατάξει των κοινοτικών διατάξεων. Ε, γίνονται ερωτήσει και οι απαντήσει είναι του τύπου δώστε μα στοιχεία ερευνούμε το θέμα το παρακολουθούμε. θέλω συγκεκριμένη απάντηση. κύριε επίτροπε έχετε την υποχρέωση να προφυλάξετε το χρήμα των φορολογούμενων τη Ευρώπη. τι θα κάνει η επιτροπή προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη πρόσωπα που βεβαιωμένα παραβίασαν την κοινοτική δομοθεσία περί προμηθειών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ναι. Στον τομέα ευθύνης μου ε, θα εμφανιστώ στο Κοινοβούλιο και στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμού για να εξηγήσω τι πρόκειται να γίνει για να εξασφαλίσουμε την καλή χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Πρόκειται για ένα ευρύτατο, για ένα σημαντικό θέμα. Άλλη μια φορά έχετε ορισμένα στοιχεία όπου ε, τα χρήματα σε έργα με συγχρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκαν ε, με λανθασμένο τρόπο, χρησιμοποιήθηκαν κακώς, ε, θα μπορούσατε να υποβάλλετε αυτές τις πληροφορίες στο τμήματά μας, θα χαρούν πάρα πολύ και θα εξετάσουν σοβαρά τα θέματα αυτά και θα εξετάσουν το ενδεχόμενο έκδοση ενός ατόμου από μία χώρα στην άλλη. Αυτό ενδιαφέρει ε, τα κράτη-μέλη και την Όλαφ και η δική, το δική μου γενική διεύθυνση δεν μπορεί να διευκολύνει τη λύση αυτή της έκδοσης για το πρόσωπο στο οποίο αναφερθήκατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση του κυρίου Μίτσελ για το λαθρεμπόριο τσιγάρων και δημόσια έσοδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ε, για αυτή τη ε, δυνατότητα που μου δίνετε να ε, τοποθετηθώ σε αυτή την ερώτηση και θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας σε αυτό το τεράστιο θέμα το οποίο πράγματι ζημιώνει τον προπολογισμό των κρατών μελών. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει, είναι ζωτική σημασία να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και η δική μας υπηρεσία, η υπηρεσία Όλαφ, ε, δραστηριοποιείται επίσης ε, ουσιαστικά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ε, του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Έχουμε μια σαφέστατη στρατηγική. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι πρώτα απ' όλα εμείς στηρίζουμε τις ε, ε, αρχές δίωξης εγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, συντονίζουμε τις δράσεις όπως ήταν την επιχείρηση «Διάβολο» Ε, που ξεκίνησε από την Κίνα. Εκεί υπήρξε λαθρεμπόριο τσιγάρων ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2008 διαπιστώθηκε ότι όλο και περισσότερο απλώνεται αυτό το πρόβλημα και η επιχείρηση Διάμπολο. Είχαμε και μία Διάμπολο 2 η οποία έλαβε χώρα το Σεπτέμβρη του 2009. Από όλα αυτά συγκεντρώνουμε πληροφορίες, τις διοχετεύουμε στους ε, εταίρους μας ε, σχετικά με τις απειλές που υπάρχουν. Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία ανάμεσα στα κρατημέλη γιατί εδώ πρόκειται για ένα θέμα που απαιτεί τη διεθνή συνεργασία. Η δουλειά της Όλαφ ε, καταδεικνύει ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία αυτή. Πρέπει όμως επίσης να σας πω ότι υπήρξαν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια των πέντε ετών ε, της Κομισιόν όπου η Όλαφ βοήθησε πάρα πολύ πρόκειται για τη συμφωνία Φίλιπ Morris και η επόμενη συμφωνία του Δεκεμβρίου 2007 ε, με την ε, μεγαλύτερη ε, επιχείρηση καπνού στην Ιαπωνία. Αυτές οι δύο τεράστιες επιχειρήσεις ομολόγησαν ότι είχαν ελλείψεις, δεν εφάρμοζαν θεμητό εμπόριο τσιγάρων και αναγκάστηκαν να καταβάλουν τεράστια ποσά πρόστιμα, τα διοχέτευσαν στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δήλωσαν ε, συνεργασία για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου τσιγάρων, κάτι που δεν τους συμφέρει προφανώς. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά εποτέγματα και αυτή η τελευταία συμφωνία καπνού με την Ιαπωνία είναι μια συμφωνία την οποία προσυπογράφουν όλα τα κράτη-μέλη. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συνεργασία σε αυτό το δύσκολο πεδίο, αλλά πιστεύουμε ότι με αυτές τις δύο μεγάλες συμφωνίες άλλαξε λιγάκι το σκηνικό και τώρα πλέον ε, διαπιστώνουμε μία έστω και μετριοπαθή πρόοδο. Όσον αφορά την περίπτωση που ανέφερε ο αξιμότιμος Ευρωβουλευτής σχετικά με την ε, παραπομπή σε δικαστήριο ενός ε, τρίτου προσώπου αυτό ε, είναι θέμα συνεργασίας Υπήρξαν αρκετέ διώξει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τα στοιχεία που έδωσε η Όλαφ. Τώρα πρόκειται για τη δίωξη ατόμου σε χώρα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο όμω εμπλέκεται άμεσα με τη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει συνεργασία σε διεθνέ επίπεδο. Μπορώ να σα αναφέρω και πολλέ πληροφορίε για συνεργασία στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Αυτό είναι θέμα που ενδιαφέρει όλους μας. Θέλουμε να ενισχυθεί η συνεργασία και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν εξαιρέσουμε το ότι ε, υπάρχει πρόβλημα με την καταγραφή, υπάρχει και πρόβλημα υγείας στο James Hotel, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ιρλανδίας, οι περισσότεροι ασθενείς έχουν ε, εισαχθεί μετά από προβλήματα λόγω του καπνίσματος. Δεν πιστεύετε ότι τελικά δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς το κόστος ε, που προκαλεί αυτό το πρόβλημα. 9,5 δις ευρώ, εξ όσων γνωρίζω, είναι ο αριθμός που αναφέρεται σε σχέση με τη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 97% αυτών δεν εντοπίζεται. Δεν έχει φτάσει πια η στιγμή η Κομισιόν να έχει μια αποτελεσματική προσέγγιση. Ίσως να εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης ε, ακτοφυλακής για να είναι περισσότερο αποτελεσματική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόσφατα επισκέφθηκα μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου επιτρέπεται το κάπνισμα. Και πραγματικά ένιωσα την έντονη διαφορά που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου δεν μυρίζει κανείς ε, πλέον ε, τον καπνό, τουλάχιστον σε δημόσιους ε, χώρους. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτό είναι το σημαντικότερο βήμα για να αποτρέψει κανείς κινδύνους στην υγεία. Όσον αφορά τώρα τον αγώνα κατά του λαθρεμπορίου. Εμείς χρησιμοποιούμε όλες τις δυνάμεις δίωξης εγκλήματος που έχουμε στη διάθεσή μας. Για μας είναι μια απόλυτη προτεραιότητα. Βεβαίως το να ε, συλλάβει κανείς, ε, να κατάσχει αυτές τις ε, ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, αυτό είναι θέμα που εμπίπτει της αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εγώ προσωπικά επισκέφθηκα ένα λιμάνι που υπάρχει μια πολύ εξελιγμένη εγκατάσταση για να εντοπίζει κανείς σκάφη που μεταφέρουν λαθρέα τσιγάρα. Αλλά σας λέω το θέμα είναι αρμοδιότητες κρατών μελών. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίξουμε διαμεσολαβητικό ρόλο, να προσφέρουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, γιατί πράγματι έχουμε πολλές δυνατότητες για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και θα συνεισφέρουμε κατά το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Όμως το να κατάσχουμε αυτό το εμπόρευμα και να το μεταφέρουμε, αυτό όπως σας είπα εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Ο κύριος Ρούμπιχ επιθυμεί να υποβάλει μια ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όσον αφορά το λαθρεμπόριο τσιγάρων, εδώ υπάρχει ε, ένα ρεύμα που χωρίζει στα τρία τα οικονομικά, το εμπόρευμα και, τα, τέλος τα παραστατικά έγγραφα. Όσον αφορά λοιπόν ε, αυτή την διακίνηση γνωρίζετε ότι θα μπορούσε κανείς ε, να επιβάλλει ένα είδος φόρου, φόρος συναλλαγής ας πούμε. Γιατί με τον τρόπο αυτό η επιβάρυνση δεν θα φορούσε ούτε το εμπόρευμα ούτε τα παραστατικά αλλά τη συναλλαγή. Νομίζω ότι για χώρες όπω με την Ελβετία αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και αξίζει τον κόπο να το σκεφτείτε. Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τις φορολογικές αρχές. Βεβαίως εμείς στην Ευρώπη... Εδώ στην Ευρώπη υπάρχει σημαντικός έμεσος φόρος κανάλωσης καπνού, γερότητα καπνικά προϊόντα και είδατε τι έγινε με τη συμφωνία Φιλιπ Μόρις για τους μεγάλους καπνοπαραγωγούς και τις ε, μεγάλες εταιρείες στην Ελβετία δεν υπήρξαν συνέπειες. Οπότε εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Όλε οι χώρε στην Ευρώπη πάντως αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα από το λαθρεμπορίο των τσιγάρων. Πάντω. ε, αν έχουμε περαιτέρω στοιχεία, βεβαίω και θα έρθουμε σε επαφή με τις ελβετικές αρχές. υπάρχει. Και άλλη μια ερώτηση που αφήνει σε εσά από τον Χάνς, Πέτερ. Μάρτιν δεν παρήσατε, επομένω θα παρελθεί αυτή η ερώτηση και πάλι σα ευχαριστούμε που ήρθατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. And now I would like to ask Mr. to take his floor. Σεύτσοβης τώρα είναι ο επόμενος επίτροπος. Υπάρχει μια ερωτήση ερωτήσεων για σας, κύριε Επίτροπε. Η πρώτη προέρχεται από την κυρία Μαρία Μπαδία Γκουτσέτ και αφορά την εκπαίδευση στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ την ερώτησή σας γιατί είναι πάρα πολύ εύστοχη και επίκαιρη. Σας τονίζω ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής Λισαβόνα για την απασχόληση επί μια σειρά ετών προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε την ανωτέρα παιδιά στην Ευρώπη. Έχουμε τρεις ε, άξονες που μας ε, απασχολούν. Η χρηματοδότηση πρώτα-πρώτα. Εδώ εφαρμόζουμε τη διαδικασία της Μπολόνια, ούτως ώστε την ανώτατη εκπαίδευση να την εξυγχρονίσουμε και να πετύχουμε στόχους μέχρι το το 2020, όπω γνωρίζετε, η διαδικασία τη Μπολόνια δεν είναι πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάτι που εντάσσεται στην διακυβερνητική συνεργασία στον τέξη ε, ευρωπαϊκών χωρών. Όμω, αναγνωρίζουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, προτέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, την υποστηρίζουμε γιατί την θεωρούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον εξυγχρονισμό τη της εκπαίδευση. Τώρα, για να σταθούμε σε κάποιε σχετικέ μα πρωτοβουλίε, περισσινές, Βοηθούμε με αυτό το τρίγωνο της γνώσης, με αυτό το Ινστιτούτο για Καινοτομία και επίσης ενθάρρυνση για κατάρτιση και παιδεία γιατί έχουμε την πρωτοβουλία για την σόβια κατάρτιση τα διπλώματα τα της επαγγελματική κατάρτισης την αναγνώριση της και κλπ. Με όλα αυτά θέλουμε η, η ανωτάτη εκπαίδευση να είναι πιο διαφανής και αντίστοιχα θέλουμε να ε, επεξεργαστούμε κάποιο είδους κατάταξη των ε, ανωτάτων ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Ο υπόψη τις ανάγκες της αγοράς απασχόλησης σήμερα και αύριο. Τι προκλήσεις αναδύονται, ιδίω για τους νέους. Αυτό το εξετάσαμε, οπότε είπαμε ότι χρειάζονται νέες δεξιότητες, νέες πρωτοβουλίες και έχουμε αυτό το επαγγελματικό και πανεπιστημιακό φόρουμ όπου ε, και επαγγελματίες αλλά και πανεπιστημιακοί ανταλλάσσουν απόψεις. Τώρα, όσον αφορά την οδότη εκπαίδευση υπάρχει συνένεση μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Έχουμε πετύχει μια σειρά πραγμάτων από το 1999 ακόμα έχει δρόμο μπροστά του αυτό το όραμα έχουμε το 2020 τουλάχιστον το 2020 και ο γύρος πλευράς διαδικασία αυτή της Μπολόνια δηλαδή στα μέσα μου χρόνια πρόκειται να επικεντρωθεί στο πώς θα βελτιώσει την κινητικότητα στην ανωτότητα εκπαίδευση πώς θα βοηθήσει την κοινωνική πτυχή πώς θα προσέξουμε την πτυχή της παγκοσμιοποίησης συνεργασία μεταξύ των ε, πανεπιστημίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε, λέει ο Πρόεδρος και τώρα. Κύριε Μπαδία, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Σήμερα, για δεύτερη φορά με ε, έχουμε τη χαρά να σα ε, υποβάλω αυτέ τις ερωτήσεις και εσείς να τις απαντάτε. Σας ευχαριστώ για όσα είπατε. Φυσικά συμφωνούμε όσον αφορά αυτή την αξιολόγηση για το τι έχει γίνει με την διαδικασία τη Μπολόνια. Όμω. Η ερώτησή μου είναι λίγο παραπέρα όσον αφορά το τι θα γίνει στο μέσο μέλλον, αλλά και ακόμα παραπέρα, πιο πολύ στο μέλλον. Γιατί τώρα μας έχει πλήξει αυτή η οικονομική κρίση, οπότε σε όλους τους τομείς και κλάδους ε, τα, τα κολέγια, τα πανεπιστήμια, τα σχολεία Πώ θα φτιάξουν νέε θέσει εργασία. Θέλουμε μια καινούργια οικονομία, την λέμε πράσινη, τη λέμε με διάφορου τρόπου. Όμω το ερώτημα είναι πώς αυτή η καινούργια κατάσταση θα, θα εξελιχθεί. Τι, τι είδους οικονομία θέλουμε να ξεκινήσει. Πώς τελειοποιηθούν όλα αυτά και τι είδους προγράμματα σπουδών θα γίνουν και στα πανεπιστήμια και στην επαγγελματική κατάρτιση. Ακριβώς σήμερα είναι η μέρα που εσείς όπως ξέρετε καλά ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία της Κοπενχάγης όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση. Παρακαλώ, πέστε μας τη γνώμη σας. Ε, Ο Επίτροπος και πάλι τονίσατε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Αυτά που σήμερα το πρωί τα συζητήσαμε, ότι τώρα έχουμε 78 εκατομμύρια που έχει εξοπλίσει με δεξιότητες η διαδικασία της Μπολόνια, outsourcing έχει γίνει, εν το του 2020 και βέβαια τώρα θα πρέπει να δούμε τι θέσει εργασία θα βρεθούν και θα πρέπει επομένω να προετοιμαστούμε. Θα πρέπει να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Για να κάτσουμε να δούμε ποιες θα είναι οι καινούργιε δεξιότητε του μέλλοντος, ποιες θα είναι οι καινούργιε δουλειέ του μέλλοντος και για τις μέλουσες και για τις νέες γενιές. Οπότε, θα συνεχίσουμε την έρευνα σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο για την κατάρτιση και την εκπαίδευση 2020 συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών. Οπότε θα συνεχιστεί η συνεργασία με όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και με τις επιχειρήσεις όσον αφορά το τι θα πετυχθεί στο μέλλον για να δούμε ποιο είναι το κατάλληλο κοκτέιλ δεξιοτήτων που θα χρειαστεί ο κόσμος του 2020. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επιτροπό για την απαντήσή του. Είναι σαφές ότι η εκπαίδευση είναι κατά κύριο λόγο θέμα των εθνικών κυβερνήσεων. Η Κομισιόν όμως μπορεί να παίξει συντονιστικό ρόλο να βάλει ένα τέρμα στο λεγόμενο εκπαιδευτικό apartheid. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχει πρόσβαση. Το δουβλένω, ας πούμε. Υπάρχουν ολόκληρες κοινότητες στον 21ο αιώνα που δεν έχουν καμία πρόσβαση στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Οι έγκλειστοι ας πούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προσφέρουμε δωρεάν εκπαίδευση σε όλους. Uh, you started your question with a very uh, clear analysis that uh, there is a division of and division of But very... Αρχίσατε την ερώτησή σας με μια πολύ σωστή ανάλυση της κατάστασης. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέκεται στο πλευρό όλων εκείνων που κάνουν κάθε προσπάθεια να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού πρόσβαση στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προσπιστούμε την ευρωπαϊκή οικονομία και την ευημερία που έχουμε στην Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη προς αυτήν την κατεύθυνση για να βελτιώσουμε και τις συνθήκες υπό τις οποίες μαθητές αλλά και σπουδαστές προερχόμενοι από μειονεκτούσες κοινωνικές ή οικονομικές ε, ε, περιοχές να έχουν πρόσβαση στην ε, ανώτατη εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Η κυρία Τιτσάου. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ υψηλό το ποσοστό των παιδιών που εγκαταλείπουν τα σχολεία. Και αν δεν επενδύσουμε επαρκώς στην εκπαίδευση και στην έρευνα θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Μόνο πέντε κράτη-μέλη επενδύουν πάνω από 2% του ΑΕΠ τους στην έρευνα και την καινοτομία. Στις άλλες χώρες και πανκοινοτικά θα έλεγα το ποσοστό αυτό ε, μειώνεται το ποσοστό δηλαδή που διοχετεύουν τα κράτη-μέλη από τον προπολογισμό τους στην έρευνα και την ε, καινοτομία αλλά και την εκπαίδευση, την παιδεία. Αυτά είναι τα μέτρα που θα πρέπει να εκρίνουν τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να υπάρχει αν μη τι άλλο ένα ελάχιστο όριο επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία και την παιδεία. Ευχαριστώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. ότι είναι εξαιρετικά υψηλό το ποσοστό των παιδιών που εγκαταλείπουν τα σχολεία. Μέχρι το 2010 θέλουμε να φτάσουμε στο 10%. Πάντως κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τα καταφέρουμε γιατί τώρα βρισκόμαστε περίπου στο 15%. Και όπως είπατε αυτό έχει πολύ κακές συνέπειες για όλους μας. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι υπό τις υπάρχουσες συνθήκες βεβαίως υπάρχουν στα δημόσια οικονομικά των κυβερνήσεων των κρατών μελών πάρα πολλά προβλήματα. η ενίσχυση των δημοσίων ε, οικονομικών ε, και οι ενέσεις ε, που προσπαθούν οι εθνικές κυβερνήσεις να κάνουν στην οικονομία είναι η πρατριότητα. Όμως όταν διέλθουμε της κρίσης θα πρέπει να κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα τονίζει με δυνατή φωνή ότι χρειάζεται να παραμείνουμε σε κατάλληλα αν μη τι άλλο επίπεδα χρηματοδότησης για πολύ σημαντικούς τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, η τεχνολογία και βεβαίως η παιδεία. Και βεβαίως οι ψηλά εργαζόμενοι σε τομείς που λένε εξελίσσονται και προσαρμόζονται στην πραγματικότητα, τη νέα κάθε φορά πραγματικότητα. Οπότε η παιδεία και εδώ έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα πρέπει να την υποστηρίξουμε ακόμα και υπό τις ε, παρούσες δυσκολίες και τους χαλεπούς καιρούς που διάγουμε. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα επίσης από την κυρία Τιτσάου πρόσβαση των νέων σε ποιοτική παιδεία αλλά και στην αγορά απασχόλησης. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι κάποια στοιχεία απάντησης έδωσα και στην προηγούμενη παρέμβασή μου. Είναι απόλυτα σαφές ότι ο τομέας αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός και θα προσπαθήσω να αναφέρω κάποια πρόσθετα στοιχεία που δεν ανέφερα προηγουμένως. Όπως ξέρετε και σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η ευθύνη για το περιεχόμενο και την ενεργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα τη ε, παιδεία και κατάρτιση. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία του θέματο που θέτει το αξιότιμο μέλος και υποστηρίζει τα μέτρα μεταρρύθμισης μέσω της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού. Το 2006 εξεδώσαμε μια σύσταση για τις ε, βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι νέοι άνθρωποι κατά την αρχική τους ε, ε, στην, στα πρώτα στάδια της προσπάθειας τους ενσωμάτωσης ε, στην ε, αγορά εργασίας. Κατά την εκπαιδευτική δηλαδή σταδιοδρομία τους. Και νομίζω ότι ε, υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να αναφέρουμε και το στρατηγικό πλαίσιο για την συνεργασία στην Ευρώπη και να τονίσουμε ότι ένας από τους ομείς προτεραιότητες στον πρώτο κύκλο αυτού του προγράμματος είναι η βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης μαθηματικών επιστημών και βεβαίως η εντατικοποίηση της προσπάθειας που πρέπει να κάνουμε για να μειώσουμε τον αριθμό των παιδιών που εγκαταλείπουν τα ε, σχολεία αλλά και των νέων που εγκαταλείπουν τα πανεπιστήμια στην ε, δυνάμει της διαδικασίας της Κοπενχάγης τα κράτη-μέλη συνεργάζονται όλο και περισσότερο και συνδυάζουν όλο και περισσότερο την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση και την αγορά απασχόληση, ώστε να βοηθήσουν του νέου να ενσωματωθούν στην αγορά απασχόληση υπό του καλύτερου δυνατού όρου. Η νέα ορμή, η νέα όθηση που δίδεται στην επαγγελματική κατάρτιση και την παιδεία είναι η βασική καινούρια ιδέα μα μέσω τη ιδέα ε, τη διαβίου μάθηση και των σχετικών πολιτικών. Είμαστε λοιπόν υπέρ μιας ε, ελαστικής αντιμετώπισης της αγοράς απασχόλησης που εξορισμού ιδιαίτερα τι μέρες μας είναι και αυτή ελαστική. Εις ό,τι αφορά το πρόγραμμα κινητικότητας Da Vinci αποδείχτηκε ένα πολύ αποτελεσματικό όργανο ε, που βοηθά τους νέους να έχουν πρόσβαση στην αγορά απασχόλησης. Αυτό αφορά κυρίως τους μαθητευόμενους, αλλά και άλλους νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά απασχόλησης. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν οι νέοι αυτοί να κάνουν κομμάτι της εκπαίδευσής τους σε άλλη χώρα και αυτό μέχρι τώρα έχει καταδείξει πολλά θετικά αποτελέσματα, βελτιώνει τις δεξιότητες ε, των ε, συμμετοχών στο πρόγραμμα, τις ε, διαπολιτισμικές τους ικανότητες, αλλά δίδει και περισσότερα του στους εργοδότες που τους προσλαμβάνουν. Ανέφερα στην προηγούμενη μου παρέμβαση το πρόγραμμα Έρασμος, αλλά στα πλαίσια των ανταλλαγών, των φοιτητών στα πανεπιστήμια. Υπάρχει όμως και μια άλλη πτυχή του προγράμματος Ερασμός που από το 2007 υποστηρίζει την εισαγωγή φοιτητών στις επιχειρήσεις. Από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό είναι, έχει επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα. 20.000 φοιτητές έχουν συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα και πάνω από 15.000 επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει σε αυτή την ε, προσπάθεια. Να, ειδού ένα παράδειγμα πώς ε, μπορούμε να αυξήσουμε την απασχολησιμότητα των πτυχιούχων, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με τον ακαδημαϊκό κόσμο και τις επιχειρήσεις. Επίσης υπάρχει και ο θετικός αντικτύπωσης της διαδικασίας της Μπολόνια για τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και των Ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Τα έχω όμως ε, πει αυτά στην προηγούμενη παρέμβασή μου, οπότε δεν θα τα επαναλάβω. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά την προσπάθεια που κάνουν να ε, ε, ενσωματωθούν στην αγορά απασχόλησης. Και βεβαίως, μην ξεχνάμε σλόγγαν της ε, προσπάθειας που γίνεται δυνάμει της στρατηγικής της Λισαβόνας More and better jobs, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Τα κράτη-μέλη δε έχουν εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Νεότητας το 2005 για να βοηθήσουν τους νέους να ενταχθούν στην αγορά απασχόλησης με ιδιαίτερα μέτρα, κάτι το οποίο βεβαίως θα είναι υποφελές προς το σύνολο της κοινωνίας. Μετά από μια πολύ φιλόδοξη και πολλά υποσχόμενη αρχή, το πρόγραμμα δυστυχώς αυτό αντιμετωπίζει, πλήττεται αν θέλετε από τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης γιατί δεν είχαμε τους πόρους που θα έπρεπε κανονικά να διοχετεύσουμε προς ε, εκεί. Και η κρίση βεβαίως ε, πρώτα απ' όλους πλήττει τους νέους, δυστυχώς. Στην ανακοίνωσή τη του 2009, δε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη και του κοινωνικού εταίρου να διασφαλίσουν ότι οι νέοι, παρά τις, ε, το δύσκολο οικονομικό κλίμα, να έχουν, να εξασφαλίσουν λίγο πρόσβαση ε, σε υψηλής ποιότητος ε, προγράμματα μαθητείας και επαγγελματική κατάρτισης και παιδείας γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιες ε, διευκρινιστικές από την κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Στην οικονομική κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε οι νέοι έχουν όλο και πιο πολλές δυσκολίες να βρουν μια δουλειά και αυτό ε, το φαινόμενο της ανεργίας δηλαδή των νέων παρατείνεται χρονικά. Μένουν στην ανεργία πολύ περισσότερο καιρό από ότι παλαιότερα. Πρέπει λοιπόν να συμμετάσχουν στον των περισσότεροι νέοι σε προγράμματα κατάρτισης ούτως ώστε να μην πληγούν ακόμα περισσότερο από τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης. Thank you. Uh, thank you. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έχετε δίκιο ότι με τις παρούσες περιστάσεις η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τις συνθήκες για τους νέους ούτω ώστε να μπορούν να κρατήσουν τις εργασίες τους ή αν τις χάσουν πώς μπορούν να επανακαταρτιστούν, να ετοιμαστούν καλύτερα για την επόμενη ευκαιρία που θα τους παρουσιαστεί για την επόμενη ενδεχόμενη απασχόληση. Η Επιτροπή εργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη και τους εμπειρογνώμονες και εστιάζονται σε τρεις τομείς. Πώς να χρησιμοποιηθεί η περίοδος αυτή, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν οι βασικές δεξιότητες και θα αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα και αρμοδιότητες. Πώς να είναι πιο δίκαιη η ανώτερη εκπαίδευση και η διδασκαλία στα σχολεία. Νομίζω ότι είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την προετοιμασία των νέων, ούτω ώστε να υπερνικήσουν τις δυσκολίες σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και να ετοιμαστούν καλύτερα για την επόμενη απασχόληση, τις επόμενες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν όταν, ε, όπως το ευχόμαστε, υποχωρήσει η κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στην ερώτηση υπαριθμών 30 που έχει ως τίτλο «Εθελοντισμό στον αθλητισμό» από τον κύριο Aylward και ίσως θέλει να απαντήσει ο Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, διότι ο εθελοντισμός ε, σε αυτές τις δραστηριότητες παίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λόγω των πλεονεκτημάτων για την κοινωνία, την συνοχή, ε, την συμπερίληψη, την ενσωμάτωση και για, τις ενδογενείς, για τα ενδογενή οικονομικά ωφέλη. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ο εθελοντισμός και ενώ υπάρχει ο αθελοντισμός σε πάρα πολλούς τομείς, υπάρχουν ε, διαρθρωτικές ε, ιδιαιτερότητες στον τομέα του αθλητισμού. Ο εθελοντισμός στον αθλητισμό είναι η βάση για την διοργάνωση, ε, διοίκηση αθλητικών δραστηριοτήτων στα κράτη-μέλη και παίζει θεμελιώδη ρόλο για την υποστήριξη του τομέα αυτού. Η σημασία του αθελοντισμού στον αθλητισμό επανειλημμένα έχει αναγνωριστεί στο πολιτικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκή ε, Βίβλο αναγνωρίστηκε ο ρόλος ε, του εθελοντισμού ως ένα από τα κοινά στοιχεία της ευρωπαϊκής προσέγγισης στον αθλητισμό. Η Λευκή Βίβλο στο πρόγραμμα δράσης, ε, υποστηρίζει τον Πιέρ του Κουμπερτά και τον εθελοντισμό στην αθλητισμό, μη κερδοφόρες δραστηριότητες και μια μελέτη για τον ενθελοντισμό και την αντιλογή βελτίστων πρακτικών. Η άτυπη ομάδα επίσης ασχολείται και με τις μη επικερδείς, μη κερδοφόρες, κερδοσκοπικές αθλητικές οργανώσεις. Μια νέα μελέτη για τον εθελοντισμό άρχισε τον, την άνοιξη του 2009 και περιγράφει τον εθελοντισμό και θα σε όλα 27 χώρες μέλη και θα έχουμε τις, την ανάλυση των διαφόρων ευκαιριών, προκλήσεων και θα ακολουθήσει η σύσταση στην, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κοινωνία των πολιτών και στις αθλητικές οργανώσεις. Η μελέτη αυτή θα περατωθεί στο τέλος του 2009 και θα τη λάβετε τις επόμενες εβδομάδες. Νομίζουμε ότι η μελέτη αυτή θα αυξήσει την κατανόηση του εθλεντισμού στον αθλητισμό και από οικονομικής απόψεως ως βάση στις απαιτήσει τις ποιοτικέ για τον αθλητισμό μέσα σε ένα πλαίσιο κοινοτικό. Όπως αναφέρεται στην πρόταση, ε, που μελετάται στην νομοθετική διαδικασία η Κομισιό προτίθεται να προωθήσει τον εθελοντισμό στην, στον αθλητισμό ε, στα πλαίσια ε, του έτους 2011 που είναι το έτος του εθελοντισμού. Εάν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, η υλοποίηση νέων διατάξεων για τον αθλητισμό θα βελτιώσει την αναφορά στην προώθηση των δομών αθλητισμού με εθελοντισμό και θα νέα σκέψη και προβληματισμό. Θα έχουμε διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους, τους ενδιαφερόμενους για να υπάρξουν δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που θα επιφέρουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ κύριος Έιλουαρντ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο και κυρίως η αναφορά του στην Λευκή Βίβλο, στον αθλητισμό. Αλλά θέλω να αναφερθώ στην παχυσαρκία που είναι από τα βασικότερα προβλήματα ε, δημοσίας υγείας. 22 ε, εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση Παιδιών είναι παχύσαρκα ε, από αυτά 4 εκατομμύρια θεωρούνται παχύσαρκα. Η αύξηση του αριθμού ε, των ε, παιδιών αυτών είναι ανησυχητική. Επίσης συνδέεται με την παχυσαρκία στους ενήλικες. Θα πρέπει κανείς να ασχοληθεί με το πρόβλημα νωρίς στη ζωή. Ή πώς θα συνδέσετε τον εθελοντισμό στον αθλητισμό με την καταπολέμηση κατά της παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, στα κράτη-μέλη. Υπάρχει κάποια δυνατότητα ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό να εισαχθεί από, τον, το δικό σας τμήμα, ούτω ώστε το, μνήμα αυτό να το μήνυμα αυτό να διαδοθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που θέσατε αυτό το σημαντικό θέμα που έχει σχέση με την επόμενη ερώτηση, αλλά συμφωνώ μαζί σας Πλήρωσω ότι η παχυσαρκία στα παιδιά και αργότερα στους ενήλικες είναι από τα πιο ανησυχητικά θέματα, είναι από τα πιο επίγοντα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αργότερα θα μιλήσω για τις μελέτες τις οποίες κάνουμε και αξιολογήσαμε σχετικά με το θέμα και είναι σαφές ότι είναι είναι δύσκολο. Από τη μια πλευρά πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να προωθήσουμε τις αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία, να τις ανθαρρύνουμε και μεταξύ των ενηλίκων και από την άλλη πλευρά να ασχοληθούμε με ε, ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, για την διατροφή. Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, είδαμε ότι στην καετία του 50 υπήρχε μεγαλύτερη πρόσληψη θερμίδων, αλλά τώρα έχουμε το πρόβλημα της παχυσαρκίας και η απάντηση είναι η σαφίσα. Ε, τότε οι άνθρωποι το περισσότερο και αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη με την παχυσαρκία μόνο με συστάσεις διαιτολογικές, διατροφικές. Πρέπει να συνδυάζεται η διατροφή με την σωματική άσκηση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σχετικά με το θέμα αυτό. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει να αποκτήσει τις αρμοδιότητες αυτές στον τομέα του αθλητισμού. Περιμένουμε να συμπληρωθεί η διαδικασία των επικυρώσεων της συνθήκης της Λισαβόνας και μετά η Επιτροπή θα αρχίσει τις διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους, τους ενδιαφερόμενους και θα προετοιμάσει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες και αυτό θα είναι σίγουρα ένα από τα θέματα πάνω στα οποία θα εστιάσουμε την προσοχή μας για να δούμε πώς μπορούμε θετικά να βελτιώσουμε την κατάσταση μεταξύ των παιδιών, να αυξήσουμε τον αριθμό των ωρών στα σχολεία που θα αφιερώνονται στην σωματική δραστηριότητα, στην φυσική αγωγή. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα αποδώσει σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάρκιν. Κύριε Επίτροπε, είπατε στην απάντησή σας ότι ο εθελοντισμός ε, συνεπάγεται ε, ξεκάθαρη οικονομική αξία και κοινωνική βέβαια. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρεται το 2011 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί η Κομισιόν προτείνει μόνο 6 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη χρονιά. Ε, το 2010 θα υπάρχει προπολογισμός 18 εκατομμυρίων. Βεβαίως ο εθελοντισμός σημαίνει ότι είναι δωρεάν, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αυτός είναι σωστός ε, λόγος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην επενδύσει σε όλους αυτούς τους εθελοντές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας για το ποσό που προβλέπετε να εκταμιευθεί για το έτος εθελοντισμού, γιατί εγώ πραγματικά πιστεύω ότι δεν επαρκεί. Ο Επίτροπος, σας ευχαριστώ πολύ ρώταγα τον διευθυντή του γραφείου μου για να μπορώ να σας δώσω μια όσο πιο ακριβή απάντηση γίνεται. Κοιτάξτε, οι πληροφορίες μου λένε ότι για το έτος εθελοντισμού 8 εκατομμύρια ευρώ θα εκταμιευθούν και νομίζω ότι με σωστό προγραμματισμό που πιστεύω ότι μπορεί να ξεκινήσει έγκαιρα από τη στιγμή που έχει ληφθεί η απόφαση ε, με σωστό προγραμματισμό και με αυτά τα χρήματα μπορούμε να προβάλλουμε τη σημασία του εθελοντισμού και το όφελος που συνεπάγεται ε, για την ε, ζωή των ε, κοινωνιών, τα ωφέλη που αποφέρει σε αυτές, ε, τα ωφέλη προς τον πολιτισμό και σε άλλους τομείς. Ελπίζω λοιπόν ότι με αυτά τα χρήματα πράγματι είναι δυνατόν, θα καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρατε στην ερώτησή σας. Επόμενη τώρα ερώτηση αφορά πάλι τον ε, αθλητισμό την ε, υποβάλλει ο κύριος ε, Κράουλη. Πρόκειται για τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η ερώτηση αυτό ε, σε κάποιο βαθμό σχετίζεται με την προηγούμενη και τις απαντήσεις που έδωσα δηλαδή πώς μπορούμε να συνδυάσουμε καλύτερες πρακτικές, πώς μπορούμε να ε, προάγουμε ένα πιο υγιή τρόπο ζωής και πώς μπορούμε να προσθέσουμε αξία σε όλους αυτούς τους τομείς. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι η Λευκή Βέβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Διατροφή, την Παχυσαρκία και συναφή θέματα, αυτή η Λευκή Βίβλος υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και η σωματική δραστηριότητα. Προτείνονται επίσης ε, δράσεις, άσκηση και ε, αυτά αναφέρονται και σε αυτή τη Λευκή Βίβλο και στη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό που και οι δύο αλληλοσυμπληρώνονται. Η Κομισιόν ε, συνέστησε μία ομάδα υψηλού επίπεδου για τη διατροφή και την σωματική άσκηση και εκεί οι εξωματούχοι από όλα τα κράτη μπορούν να έχουν έτσι μία γενική εικόνα για τις ε, πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις στον τομέα αυτό. Όπως γνωρίζετε αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου ε, πρόκειται να συναντιέται τρεις φορές το χρόνο. Μέσα από το πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας η Κομισιόν έχει στηρίξει μεταξύ άλλων πρωτοβουλίες ε, που έχουν ως στόχο τη διατροφή και τη σωματική άσκηση κυρίως των νέων. Επανέρχομαι στη Λευκή Βίβλο για τη διατροφή. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσω ότι το έγγραφο αυτό υπογραμμίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας και η ΜΚΟ καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο να μας βοηθήσουν να διασφαλίσουμε ότι πράγματι θα μειωθεί η παχυσαρκία. Όσον αφορά τώρα τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τη διατροφή τη σωματική άσκηση, αυτή η δουλειά συνεχίζεται και τα μέλη της πλατφόρμας καλούν ε, να υπάρξει δραστηριοποίηση. Στον τομέα του αθλητισμού η Λευκή Βίβλος παραμένει το μόνο σημαντικότερο σημείο αναφοράς και προβλέπει διάφορες δράσεις στον τομέα του αθλητισμού και της υγείας. Όλα αυτά είναι γνωστά κάτω από τον τίτλο «Δραστηριότητες που ενισχύουν την υγεία». Και εδώ συμπεριλαμβάνεται και το δίκτυο του ε, HPA. Εξάλλου προβλέπονται περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης σε αυτό τον τομέα, παρήματος χάρη στο πλαίσιο του 7ου προγράμματο δράση για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, ε, το ε, πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη διαβίου μάθηση και πολλά άλλα. Οι ε, κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σωματική δραστηριότητα που εγκρίθηκαν το 2008 μπορούν επίσης να εκλειφθούν ως μια συνεισφορά σε ενημερωμένους πολίτες για τα ωφέλη της ε, σωματικής δραστηριότητας έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή εφαρμόζει, αναλαμβάνει δράση στον τομέα του αθλητισμού έτσι ώστε και στο μέλλον υπάρχουν δράσεις ε, με βάση τις ε, αποφάσεις προπολογισμού που πήρε το Κοινοβούλιο και οι ε, προκατακτικές δράσεις του 2009 έχουν ήδη δείξει πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στον τομέα αυτό, όπου το 64% των αιτήσεων αφορούν ακριβώς την υγεία και τη διατροφή. Ευχαριστώ. Mr. Crowley. Ευχαριστούμε. Κύριε Κράουλη, θέλετε το λόγο. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τόσα απήντησε. Όμως είπατε κάτι παραπάνω, γιατί θα πω δύο πράγματα. Πρώτα πρώτα για αυτή την ομάδα σε σχέση με την διατροφή. Όμως έχουμε και τις προβληματικές διαφημίσεις. Κάθονται και λένε ότι ο αθλητισμός σχετίζεται με κάποια προϊόντα, κάποια πρόσθετα. Όμως αυτό οδηγεί σε βλάβες της υγείας. Γιατί χρησιμοποιούν αυτές τις ορμόνες. Διάφορα ποτά για καλύτερες επιδόσεις και θεωρούν ότι έτσι θα έχουν έξτρα απόδοση. Αυτό όμως οδηγεί σε προβλήματα υγείας. Το θέμα είναι να ενθαρρύνουμε και τον κοινό άνθρωπο και, και τους αθλητές ότι τέτοιου προϊόντα δεν είναι εδώ να τους κάνουν ποτέ προαθλητές. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Επίτροπος, ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι πάρα πολύ εύστοχα το είδατε το πράγμα. Στο οποίο παιδιμαστήριο θα δει κανένα ε, ολόκληρα ράφια γεμάτα με διάφορα τέτοια προϊόντα. Και πρόσθετα διατροφή. Ολόκληρη βιομηχανία έχει στηθεί Νομίζω ότι έχετε δίκιο 100%. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να κάτσουμε να προβληματιστούμε. Να βρούμε την κατάλληλη προσέγγιση, να βρούμε την πιο ισορροπημένη λύση, τόσο ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο που κάνει σπορ τη δυνατότητα να διαλέξει προϊόντα, να έχει τη σωστή πληροφόρηση σε σχέση με το τι προϊόντα καταναλώνει. Άρα χρειάζεται μια εκστρατεία ενημερωτική όσον αφορά τις συνέπειες τέτοιων πραγμάτων και προϊόντων. Βέβαια και από πλευρά προστασία του καταναλωτή θα πρέπει να περιγράφονται αυτά τα προϊόντα, θα πρέπει να είναι γνωστό ποιε είναι δυσμενεί συνέπειε που η κατανάλωση τέτοιων προϊόντων είναι δυνατόν να έχει για του αθλωμένου. Άρα έχετε δίκιο 100%. πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε πώ μπορούμε να αποκλείσουμε τι αρνητικέ συνέπειε. Μην κάνουμε δηλαδή αθλητισμό και μετά ε, ανατρέπουμε τι ε, θετικέ συνέπειε με αυτά τα βλαβερά προϊόντα. Ο πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Η τελευταία ερώτηση, κύριε Επιτροπή, για σας, για απόψε. Ο κ. Κάτσιν έχει υποβάλει την και αφορά τις δυσκολίες για το σλοβένικο θέατρο της, ε, της, της, της, της της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να κάτσουμε και να πρέπει να βρούμε τι γίνεται. Πώς να βοηθήσουμε το θέατρο αυτό, πώς να βελτιώσουμε την κατάσταση για αυτό το θέατρο. Ξεκινώ τονίζοντά σα ότι όσον αφορά την κοινωνική δράση έχουμε το άρθρο 151 το οποίο προβλέπει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει τη συνεργασία των κρατών μελών και αν χρειάζεται να δράσει συμπληρωματικά. Παρ' αυτά. Η ταμεία ειδικών πόρων για αυτά τα ιδρύματα είναι θέμα κρατικό. Δεν παίζει εδώ κοινωτική αρμοδιότητα. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο πολιτιστικό διάλογος αλλά και η προώθηση της πολυμορφίας πολιτικής είναι στόχος κλειδί. Και κάποια διακριτικά projects, επομένω, είναι δυνατόν να επιλέξουμε τόσο ώστε να υπάρχει στήριξη από πλευρά κοινότητα σύμφωνα με κάποια πολιτιστικά προγράμματα. Άρα, πιο συγκεκριμένα, θέλουμε να φέρουμε την ε, δημιουργικότητα, την κινητικότητα των καλλιτεχνών, την προσβασιμότητα του κοινού, την διάδοση της τέχνης, αλλά και το διαπολιτιστικό διάλογο, αλλά ταυτόχρονα την γνώση της πολιτικής ιστορίας των λαών της Ευρώπης. Και μόνο κάποια τέτοια προγράμματα με ευρωπαϊκή διάθεση είναι δυνατόν να καλυφθούν. Και χρειάζονται κάποια μήνυμα Όσον αφορά το πόσοι, πόσα κράτη που συμμετέχουν τώρα, οι ενισχύσει μονοδιάστατων projects γίνονται μόνο αν έχουμε 700 που συμμετέχουν. Επίσης, εμείς έχουμε εκπονήσει μια στρατηγική ούτως ώστε να προαγάγουμε την πολυγλωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό καλύπτει επίσημε, εθνικέ, ε, μειονοτικές γλώσσε, γλώσσε των ε, μεταναστών. Το συνέδριο 2008 προέβηνε κάποια σχετική ανακοίνωση και δεσμευτήκαμε ώστε να καταστεί βέβαιο ότι είμαστε υπέρ όλων των γλωσσών που μιλούνται στην ευρωπαϊκή κοινότητα και των γλωσσών των μειονοτικών. Έχουμε κάποιε στρατηγικέ οι οποίε ε, υλοποιούνται σε στενή εργασία με τα μέλη, οπότε τελικά τα κράτη-μέλη θα πρέπει, όσον αφορά την ιστορική γλωσσική πολιτική, να λάβουν τι αποφάσει. Η ιδέα προαγωγή της, ε, των γλωσσικών ε, καταρτήσεων και γνώσεων είναι ένας από τους στόχου του προγράμματος για την σοφή κατάρτιση. Το ίδιο αφορά και τα προγράμματα για τον αθλητισμό, τα δίκτυα, ούτω ώστε έτσι να βοηθούν όλε οι γλώσσε και οι μειονοτικέ Πέραν αυτών. Σας τονίζω ότι προστασία των μειονοτήτων είναι βασική ιδρυτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένω θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα νομικά μέσα ούτως ώστε να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα και των μειονοτήτων και επίση αποφασιστικά να δρώνουν κατά ή ασδήποτε διάκριση. Ευχαριστώ. Εσείς κύριε Κάτσιν θέλετε να προβείτε σε η ερώτηση. Μάλιστα. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για το όσο μας απαντήσατε. Καταρχήν, απαντήθηκε η ερώτησή μου, όμως δεν νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Είναι σημειακό, πολύ συγκεκριμένο, διότι θεωρείται ότι αυτά τα θέματα είναι εθνική αρμοδιότητα. Όμως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι κάποια θέματα δεν τα χειρίζεται σωστά η Ιταλία και γι' αυτό και κάτσαμε και φτιάξαμε ένα ψήφισμα το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει τα δρόμενα στην Ιταλία. Εσείς θεωρείτε όμως ότι δεν υπάρχει νοτική αρμοδιότητα. Η πλειοψηφία εξημών όμως θεωρεί ότι θα έπρεπε εσείς να εμπλακείτε επίσης σε αυτό το θέμα γιατί το θέμα της μειονότητας δεν είναι μόνο θέμα δικαιωμάτων πολιτών, είναι και θέμα υποχρεώσεων είναι υποχρέωση του κράτους να προστατεύσει τις μειονότητες. Χαίρομαι που μιλήσατε για δυσμενείς διακρίσεις και για την καταπολέμηση του φαινομένου. Όμως, δεν είναι το να επιβιώσει καμία μειοψηφία εκτός εάν υπάρχει θετική διάκριση. Αυτό χρειάζονται οι μειονότητες. Ηθική, οικονομική στήριξη για να επιβιώσει. Θετική διάκριση. το θεσμικό μας όργανο συγκροτήθηκε εδώ και 50 χρόνια και έτσι και λειτουργεί. Όμως, κάθε χρόνο έχουμε την ίδια ιστορία. Για όλους όσους δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, ουσιαστικά τους ασκείται πολιτική πίεση. Επομένω, αυτό στη συγκεκριμένη, τα συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα είναι, είναι ο όρο προπόθεση επιβίωση. Ευχαριστώ, Επίτροπο. Καταλαβαίνω 100% αυτά που σα ταλανίζουν. Όμω, εμεί στην Κομισιόν πρέπει να λειτουργήσουμε βάσει κάποιων κανόνων οι οποίοι έχουν θεσπιστεί, ιδίω όσον αφορά την εκταμίευση των πόρων. Οπότε και στην απάντησή μου προσπάθησα να σας εξηγήσω ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε σε, από Ευρώπη Ευρώπης για να κάνουμε κάτι για το σλοβενικό θέατρο. Ο μόνος τρόπος που κάτι μπορεί να γίνει είναι να υπάρχει συνεργασία και έτσι να υπάρχει ενεργή συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα υπό τι σημερινέ προποθέσει. Αυτό είναι εφικτό και θα ωφελήσει και αυτό το θέατρο και άλλους που τυχόν θα συνεργαστούν στο μέλλον. Μόνο από αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θετικά να κάνει κάποιες κινήσεις. Κάτσε και να αξιολογήσει αυτή την ευρωπαϊκή συνεργασία. Όπως ξέρετε δεν υπάρχει κονδύλιο το μπορεί να προβλέπετε για τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές είναι φορτισμένη συζήτηση για τέτοια θέματα. Γιατί σας απασχολεί. Είναι θέμα εθνικότητας, είναι θέμα γλώσσας. Οπότε το κοινοβούλιο είναι αυτό το, το, το, το κατάλληλο όργανο για να συζητηθούν τέτοια πράγματα, όπως είπα και στην συμπληρωματική ερώτηση. Ξαναδεύτε τέλειωσε των ερωτήσεων. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε. Και περιμένω πώς και πώς να τα ξαναπούμε.